του Νοεμβρίου 2009. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την έκθεση Μπέγκε. Είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία, είναι ονομαστική κλίση. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Μπέγκε. Προχωράμε στην έκθεση της κυρίας Ματέρα σχετικά με την κοινοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου What is this? Okay. Ο κύριος Χάρτον επί της διαδικασίας, παρακαλώ. van Nederland. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ντόλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ψήφισε για το 6% την αύξηση ε, του ε, ευρωπαϊκού προϋπολογισμού εις βάρος των ευρωπαίων φορολογουμένων. Ε, η δική μου ομάδα και το κόμμα μου είναι κατηγορηματικά αντίθετη και προσβάλλεται και τη χώρα μου με αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε και έχει κλείσει η συζήτηση. Προχωράμε. Mr. President. Mr. Doe, go ahead. Yes, please. Oui, mes chers collègues. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Αποφασίσαμε στην τελευταία διάσκεψη των Προέδρων να εγγράψουμε σημερινή ημερήσια διάταξη στην έκθεση Ματέρα. Ουδής ε, ζήτησε να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη το μόνο που απασχολεί τον πρόεδρο είναι αν θα κάνουμε τέτοια συζητήσεις ειλικρινής απέναντι ε, ε, σε τέτοια άτομα όπως αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Ε, συζητήσεις που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πέντε χρόνια. Εάν στέλνει η ομάδα του αυτό τον κύριο στη διάσκεψη των Προέδρων πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία της ε, πρώτης έκθεσης της κυρίας ε, Ματέρα ε, για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι η κυρία Ματέρα είχε ζητήσει το λόγο, αυτό ισχύει, ως δραπορτέρ ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε κληθεί να ψηφίσουμε ένα πακέτο βοήθειας υπέρ της Ολλανδίας που ζήτησε κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για ένα συνολικό ποσό της τάξης των 10.500.000 ευρώ. Αυτή η μεταφορά κονδυλίων εντός του προπολογισμού θα τηρήσει την συνήθη πορεία, αλλά οι επόμενες αιτήσει βοήθειας που αυξάνονται συνεχώς, μπορεί και να σταματήσουν λόγω της μη έγκρισης ακόμα του προπολογισμού του 2011. Εάν το σύστημα των 12 ξεκινήσει να ισχύει από τον Ιανουάριο, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις μεταφορές και να προχωρήσουμε με τις κατάλληλες πληρωμές. Και επειδή ακριβώ βιώνουμε δύσκολη οικονομική κατάσταση για όλη την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξει ένα μεγάλο αίσθημα ευθύνη, όπω το ίδιο περιμένει και από τα κράτη-μέλη που ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου ε, εξέφρασαν ενστάσει για την ε, έγκριση και ε, αυτά όλα είναι, υπέρ της, είναι και βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ονομαστική, ψήφο η, η έκθεση κυρία Ματέρα για το Ινστιτούτ Όλαντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, η ημερήσια διάλυση προβλέπει την επόμενη έκθεση της Ματέρα, πάλι για το Globalization Adjustment Fund, ε, στο Δρένθε, κλάδο κλάδος 18, από τις κάτω χώρες. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση πάλι της κυρίας ε, Ματέρα για το Ταμείο Προσαρμογής Παγκοσμιοποίηση η αίτηση για το Λίμποργκ. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η επόμενη έκθεση πάλι της κυρίας Ματέρα ε, για το Ταμείο Προσαρμογής Γκάλτερλαντ και Όβρισελ με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ε, επόμενη έκθεση της κυρίας Ματέρα πάλι. Ταμείο Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση. Νουρτ Χόλαντ ε, και Ούτρεκτ. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση της κυρίας Ματέρα για Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νουρτ Χόλαντ και Ζουτ Χόλαντ με ναι, ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Ματέρα. Η μερίσια διάθεση προβλέπει ψηφοφορία ε, επί της έκθεσης του κυρίου Ντεκάστρο σχετικά με ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του γερμανικού μονοπωλίου αλκοόλης με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντεκάστρο. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση της, ε, του κυρίου Μορέιρα σχετικά με τη δασμολογική ατέλεια για συγκεκριμένα φαρμακευτικά δραστικά συστατικά που φέρουν διεθνή κοινή ομονομασία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Μορέιρα. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση του κυρίου Ρεούλ σχετικά με την ανανέωση της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ουκρανίας. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται η επόμενη έκθεση πάλι του κυρίου Ρεούλ σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας Επιστημονικής Τεχνολογικής Συνεργασίας ε, μεταξύ της ΕΕ και της κυβέρνησης των νησών των, των Φερόε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η έκθεση του κυρίου Ρεούλ ε, για τη σύναψη παρόμοιας συμφωνίας με την κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη έκθεση αντίστοιχη συμφωνία με το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Ρεούλ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει φοφορία από τις έκθεσης της κυρίας Πατράου Νέβες σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας αλλιευτικής σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νήσων του Σολομόντος. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια η επόμενη έκθεση του κυρίου Κάζα σχετικά με κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Η επόμενη έκθεση, η έκθεση του κυρίου Μπάλτς σχετικά με την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2009. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση του κυρίου Έλλερ σχετικά με την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικοστρατιωτικών ικανοτήτων. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Μπιλμπάου Μπαραντίκα σχετικά με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση του αποθέματος γάβρου. ...το βυσκαϊκό κόλπο και τις ελιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος. Η εισηγήτρια ζητάει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θα ήθελα να πω ότι στην Επιτροπή Αλίας καταψήφισε την έκθεση γιατί ορισμένες τροπολογίες που είχαμε επεξεργαστεί με τους αλείς δεν έγιναν δεκτές. Πάντως το πιο σημαντικό για μένα είναι να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο τέτοιο σχέδιο διαχείρισης του γαύρου. Γι' αυτό και τώρα θα υπερψηφίσω και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο που είχε σοβαρού συνδυασμού και επιφυλάξει να δεχθεί την ικανότητα συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπω κατοχυρώνεται με τη συνθήκη τη Λισαβόνα και σας παρακαλώ από σήμερα να θέσετε μια ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, γιατί ο ληφτικός κλάδος ε, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση αν δεν προωθηθεί αυτό το σχέδιο και δεν εφαρμοστεί. Τροπολογίες της Επιτροπής 1 με 36. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Ε, η πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με ονομαστική κλίση το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Μπιλμπάου. Η μερίσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία τη έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ σχετικά με τη θέσπιση πολιετού σχεδίου για το δυτικό απόθεμα Σαφριδιού και για την αλληλεία του αποθέματο αυτού. Ψηφίζουμε πρώτα σε μία σειρά από τροπολογίες της Επιτροπής 1, 8, 10, 19, 21, 28. Ο ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τροπολογία 29 αποσύρθηκε από τους σοσιαλιστές για λόγους που μου διαφεύγουν για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, σας διαβεβαιώ ότι θα προχωρήσουμε με αυτή την τροπολογία. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα ήθελα να το σκεφτούν τα μέλη κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πλήρως το νόημα αυτού του πράγματος. Τι κάνουμε αν δεν δεχτούμε την τροπολογία των σοσιαλιστών και δεχτούμε την ε, τροπολογία του ΕΛΚ σημαίνει ότι αντιβαίνουμε στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και δημιουργούμε δύο διαφορετικές ε, περιοχές ε, για τα επιτρεβόμενα αλλιεύματα. Ε, προτείνω λοιπόν να καταψηφίσουμε την τροπολογία του ΕΛΚ και να εγκρίνουμε την ε, ε έκθεση των σοσιαλιστών παρά το γεγονό ότι την επέσυραν. Ε, έχει γίνει για πολύ σοβαρούς λόγου για τα νότια τμήματα τη Ευρώπη. Με άλλα λόγα κύριε Γκάλαγκερ, επικαλείστε τον κανόνα 156 σημείο 5 και εγκρίνετε την τροπολογία 29 και δέχεστε να περάσει στο κατάλογο των ψηφοφοριών, επομένω πρέπει να την ψηφίσουμε. Τροπολογίες 1, 8, 10, 19, 21, 28. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Α, τροπολογία 30 και 31. Ταυτόσιμες. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Α, Let's check. Let's Τροπολογίες 30 και 31. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Επομένως, καταπίπτει η 9, καταπίπτει η 29 και ψηφίζουμε την ε, πρόταση όσους τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Κάλαχερ. Η μερίσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Γκρόμπερτσικ σχετικά με την απαγόρευση διαλογής αλλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας και τους περιορισμούς αλληλείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι στα ύδατα της Βαλτικής θάλασσας, των Μπέλτς και του Σάουντ. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η πρόταση ως τροποποιήθη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Έκθεση του κυρίου Ζωάου Φερέιρα σχετικά με τη χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξενικών και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα ως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Ναι. Το ψήφισμα ως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε στις 12 η ώρα μιλάει στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Γεωργίας. Θα προχωρήσω στην ψήφου επί της έκθεσης ΡΑΠΚΑΙ. Μετά θα διακόψω για την ομιλία και θα συνεχίσουμε τις δύο εναπομείνουσες ψηφοφορίες, είναι μικρές, μετά την ομιλία του Πρόεδρου Γεωργίας. Προχωράμε, προχωράμε, thank you for your approval. Σας ευχαριστώ για την έγκριση που δίνετε στην πρότασή μου. Το εκτιμώ Έκθεση ΡΑΠΚΑΙ. Ε, μία σειρά από τροπολογίες της Επιτροπής, μία έντεκα κτλ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. No, I will not. Or I will if you want me to waste time. Όχι, δεν θα το κάνω, εκτός και αν θέλετε να χάσουμε χρόνο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα οφορίας. Εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 33 και 31 καταπίπτουν. Τροπολογία 39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 27 καταπίπτει τροπολογία 28 με ονομαστική κλίση Άρκετη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία 34 καταπίπτει. Τροπολογία 35. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. I Θα κάνω έλεγχο για να χάσουμε λίγο χρόνο. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγώ λέω ότι απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Check. Πέρας προφορίας. And it is απορρίπτεται. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 καταπίπτει. Τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 31 καταπίπτει. Τροπολογία 32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Okay, this is fun. 32. I said εγκρίνεται. Check. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται με ονομαστική κλίση το ψήφισμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Ράπκαη We will now break the session the... Θα διακόψουμε τώρα για την ομιλία του Πρόεδρου της Γεωργίας και θα συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες και τις επεξηγήσεις ψήφων μετά το πέρας της ομιλίας.